λόγο στον κύριο Γερσί Μπούζεκ. Έχετε το λόγο κύριε Μπούζεκ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Αγαπητέ αντιπρόεδρε, έχουμε και αλλαγή τώρα σκητάλης όσον αφορά την ε, ε, προεδρία. Υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό για να προαχθεί η ευρωπαϊκή οικονομία με τα δεδομένα και πρέπει να είναι φιλόδοξη σε σχέση με τα μέγα δεδομένα big data η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και να προστατεύει τις αξίες μας πρώτα απ' όλα τον ιδιωτικό χαρακτήρα τον χαρακτήρα του απόρριτου αυτών των στοιχείων θα πρέπει να δημιουργήσει μια βάση, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο η Ευρώπη ώστε να μπορέσει να προαχθεί η ασφάλεια των δεδομένων και ιδιαίτερα να προαθεί η ιδιωτική επένδυση όσον αφορά τις υποδομές, την έρευνα και την ανάπτυξη. Τρίτη παρατήρηση να δημιουργηθεί μια αυθεντική ψηφιακή ένωση με την προστασία πνευματικών και συγγενών δικαιωμάτων, τέταρτος άξονας, να μπορέσουν οι εταιρείες που ξεκινούν την δραστηριότητά τους, startups, να ενισχυθούν, να υποστηριχθούν και να εμπλακεί η κοινωνία πέμπτος άξονας ώστε να επωφεληθεί από τα μέγα δεδομένα και να υπάρξει η μέγιστη, βέλτιστη χρήση τους. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει παγκόσμιος διεθνής προπομπός, πρωτοπόρος Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για την συνεργασία στο επίπεδο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, για την προαγωγή αυτού του ζητήματος ε, των δεδομένων. Και να πω ότι αμέλησα την αναφορά ενό πολύ σημαντικού θέματος στην προστασία των καταναλωτών και των δικαιωμάτων των καταναλωτών θα πρέπει εδώ σε σχέση με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή να ληφθούν υπόψη αυτές οι παρατηρήσεις και εσείς να τις λάβετε υπόψη, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Thank much, uh, Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Φόρντ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. Ο ψηφιακός κόσμος δεν γνωρίζει σύνορα και δημιουργούνται νέα ερωτηματικά λόγω των και πρέπει να συνεργαστούμε όλοι, με όλους. Τα μαζικά δεδομένα ε, διευκολύνουν ε, τις πωλήσει των επιχειρήσεων, ε, τη μείωση του κόστου, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, έχουν ρόλο κλειδί για την ανάπτυξη της οικονομίας. Όμως το ρυθμιστικό περιβάλλον θα πρέπει να λειτουργεί σωστά και για τους καταναλωτές, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις. Μπορούμε να έχουμε σημαντικά ωφέλη. Πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές ε, και φυσικά θα πρέπει ισχύουν και ισότιμη ώρα ανταγωνισμού, το οποίο ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων καθώς και την κοινοτομία. Ε, νέοι τομείς, ε, όπως παραδείγματος χάρη οι μεσίδες ε, των βασικών δεδομένων, δημιουργούν νέα ζητήματα, όπως αυτό της διαφάνειας. τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρακολουθεί αυτούς τους νέους τομείς και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια ψηφιακή ουδετερότητα για να μην διονίζονται παλιά μονοπόλια, ε, νέα φάρμακα, νέοι τρόποι προστασίας του περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας, αποτελεσματικότερες δημόσιες υπηρεσίες. Ε, ανοίγονται νέες πόρτες, όμως ε, θα πρέπει να ξεκλειδώσουμε αυτήν την νέα ευφυή τεχνολογία. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να υπάρξει ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και να επιτρέψει κρατικέ προμήθειες που βασίζονται σε νέε τεχνολογίες ήδη το περασμένο καλοκαίρι υπέβαλε αυτή την ερώτηση και καταλήξαμε να το συζητούμε τώρα το Μάρτιο. Πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα. Ε, έχουμε ε, ε, καλά νέα για την προστασία των δεδομένων πέρα, όμως από την Ευρωπαϊκή Φυσαλίδα μην ξεχνάμε ότι συμβαίνουν πράγματα. Ο Ευρωπαίος επόπτης των δεδομένων είναι υπερβολικά προσεκτικός και έτσι βάζει ένα ζουρλομανδία γύρω από τα δεδομένα δεδομένα και ασφικτιούν. Θα πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα στην ευφυή τεχνολογία. Χρειάζεται σωστή καθοδήγηση για να χρησιμοποιήσουμε τα μαζικά δεδομένα για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές, για τους ερευνητέ και τους παρόχους υπηρεσιών. Ε, χρειαζόμαστε νέες καθαρές τεχνολογίες. Αυτό είναι ένα βήμα, όμως χρειαζόμαστε τώρα υλοποίηση και ξεκάθαρες κυρίως κατευθυντές γραμμές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Φόρντ. Ο Αντιπρόεδρο Άνσιπ έχει το λόγο, ο εξονόμος Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, Σα ευχαριστώ για τι ερωτήσει που συζητούμε σήμερα. Δείχνουν ότι και η ώρα για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι δυνατότητε που παρέχει η ψηφιακή οικονομία. Η οικονομία των δεδομένων αναπτύσσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα φτάσει τουλάχιστον το 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. Πρέπει να γίνει ακρογωνίως λίθος της οικονομίας μας, να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, υπηρεσίες και νέα επιχειρηματικά πρότυπα. Στις πρόσφατες διαβουλεύσεις της δημόσιας, θέλαμε να ανταλλάξουμε απόψεις για να κατανοηθεί ο ρόλος ε, της αγοράς δεδομένων, της πρόσβασης δεδομένα και της ελεύθερης ροής δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χαρτογραφήσει, χαρτογραφεί συγγνώμη, τους περιορισμούς ελεύθερης ροής των δεδομένων και θα αξιολογήσει τα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά την πρόσθεση των επιχειρήσεων στα δεδομένα και πώς θα γίνεται η χρήση και εκ νέου χρήση των ε, δεδομένων και ε, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των μη προσωπικών δεδομένων. Είναι το νέο πετρέλαιο τα δεδομένα. Χρειάζεται διαλειτουργικότητα, χρειάζονται προδιαγραφές. Και αυτή είναι η αγωγή για τα δεδομένα επεξεργαζόμεθα προτεραιότητες για την τυποποίηση των δεδομένων και τη συναφείς δράσεις σε βασικούς τομείς τεχνολογίας για να έχουμε μια ψηφιακή ενή αγορά η οποία μπορεί να οδηγήσει στη σωστή τυποποίηση. Όσον αφορά το νέφος θα υιοθετήσουμε ε, τη χρήση του υπολογιστικού νέφου στου τομεί που θεωρούμε ότι είναι υποφελέ για την παραγωγικότητα. Για να ψηφιοποιήσουμε της ε, δημόσιας δικήσης. θέλουμε στα πλαίσια της ενιαίας ψηφιακής αγοράς να έχουμε μια νέα, ένα νέο σχέδιο για ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σύμφωνα το σχέδιο δράσεως έχω στόχο την επιτάχυνση της εφαρμογής ανοιχτών και ενωτόμων και συνεργασίμων κυβερνήσεων που θα υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα και τις διασυνοριακές ε, δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες. Χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό ε, κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων. Χρειαζόμαστε και αναθεώρηση των κανόνων περί προστασίας ιδιωτικής ζωής και προστασία του κυβερνοχώρου και των ε, καταναλωτών. Και έτσι θα υπάρχει εμπιστοσύνη όσον αφορά την οικονομία των δεδομένων. Θέλουμε να αυξήσουμε την ασφάλεια δικαίου. Θέλουμε να έχουμε ομοιόμορφους κανόνες. Έτσι θα εγγυόμεθα ισότιμες συνθήκες της επιχείρησης. Θα μπορούν να ανταγωνίζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση όρης. Η συγκεκριμένη κατάσταση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει ληφθεί υπόψη. Και έχουμε κάνει προτάσεις για τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσεξε να μην αυξήσει το διοικητικό άχθος τη μικρομεσαίες επιχειρήση. Οι επιχειρήσεις αυτές θα ωφεληθούν από προστευμένο κανονιστικό περιβάλλον που παρέχει ο κανονισμός και ο μηχανισμός ενιαίας θηρίδας των εθνικών εποπτικών αρχών θα βοηθήσει επίσης. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τα δεδομένα όμως. Χρειάζονται σωστέ δεξιότητε και ικανότητε για την επεξεργασία των δεδομένων με σωστό τρόπο και να δημιουργηθούν νέε επιχειρήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει θεματολόγιο για τι δεξιότητε για την Ευρώπη στο πρόγραμμα εργασιών του 2016. Θέλουμε να προωθήσουμε τι δεξιότητε Θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες που μπορούν να δημιουργηθούν για ψηφιακές θέσεις απασχόλησης. Σε μια ερώτηση ετέθη το θέμα α, του μπορεί των δεδομένων, αν θέλετε. Παρακολουθούμε το σύγνεγγις, τη δημιουργία αυτών των αγορών δεδομένων. Θέλουμε να αξιολογήσουμε αν χρειάζεται δράση και πολιτική. Για να γίνει αυτό πρέπει να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς που δημιουργούνται. Πρέπει να βρούμε τη σωστή τιμή και σύνθεση των δεδομένων προς εμπόριο ε, και πώς επηρεάζεται η οικονομία ψηφιακή. Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη διαφάνεια, στον έλεγχο και στην αμεροληψία. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Ξεκινάει η συζήτηση για τις πολιτικές ομάδες. Συνάδελφε Μπόνη, έχετε το λόγο 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, Ποιος είναι... Ποιος είναι ο στόχος ε, για το ότι μια οικονομία με βάση τα δεδομένα μπορεί να δώσει πιο αποτελεσματικά προϊόντα, πιο φιλικές υπηρεσίες για τους χρήστες και ατομικές ε, λύσεις. Μπορούμε να πούμε ότι τα δεδομένα με την επιστήμη με τις πόλεις, ευφυείς πόλεις, smart cities που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά. Επίσης για την δράση στον τομέα της υγείας και με την επικοινωνία σε σχέση με ε, ρομπότ και ανθρώπους ώστε να έχουμε αποτελέσματα προς όφελος όλων. Είναι η μοχλευτική αυτή αποτελεσματικότητα που μπορεί να συνεισφέρει ώστε να αναβαθμιστούν οι επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο, ρυθμιστικό και μη. Νέες τεχνολογίες που απαιτούν περισσότερο ήπιο δίκαιο, ήπιου χαρακτήρα ρυθμίσεις ε, όσον αφορά και την ε, ασφάλεια και τα προσωπικά δεδομένα αλλά και την καλύτερη χρήση τους για να επιληθεί το πρόβλημα της ιδιοκτησίας, της κυριότητας των δεδομένων. Ανοιχτά δεδομένα στην προσπελασιμότητα με την δυνατότητα να χρησιμοποιούνται για δημόσιους σκοπούς και υπηρεσίες. Ε, η πέμπτη γενεά να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από αυτά τα δεδομένα για τις ε, ε, δυνατότητες υψηλών επιδόσεων ε, υπολογιστών και νέφους. Η κάλυψη των διαλειτουργικών δυνατοτήτων πανευρωπαϊκά. Όλα αυτά σαν σύνολο δημιουργούν ε, νέες ευκαιρίες ε, για την δράση μας. Δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε. Αναμένουμε λοιπόν συνεκτικές και συναφείς προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα είναι αποτελεσματικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από την ίδια πολιτική ομάδα δεν μπορούμε να δεχτούμε γαλάζια κάρτα. Ε, η κυρία σας ευχαριστώ. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Θέλουμε να ανθίσει, να γίνει πιο ανταγωνιστική. Και μπορούμε να έχουμε μεγάλη ευκαιρία με την οικονομία των δεδομένων. Ξέρουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί αυτομάτως και αυθορμήτως. Θα πρέπει να είναι καρπός ευρωπαϊκής στρατηγικής. Δεν θα συμβεί ως εκθαύματος και αυθορμήτως. Έχουμε πολύ δρόμο να καλύψουμε, διότι ξέρουμε ότι οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει πολύ, ξέρουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι big σε αυτή την οικονομία του big data. Ίσως μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να κάνει πολλά πράγματα ακόμα. Επενδύσεις, όπως υπόθηκε. Χρειάζεται διαλειτουργικότητα, διότι μηχανήματα και αισθητήρε πρέπει να συνεννοούνται μεταξύ τους θα πρέπει να συμμετάχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι εταιρείε για τη χρήση. Χρειάζονται ε, μεγαλύτερη επικοινωνία. Πρέπει να κάνουμε πολλά. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να δούμε και μακρόπνα τα πράγματα. Το είπε ο πρόεδρο Μπούζεκ. Πρέπει να κοιτάει μπροστά η Ευρώπη, να είναι καινοτόμα, αλλά να υπερασπίζεται τι αξίε τη, να τι παγιώνει. Χρειάζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα στρέφεται προ το μέλλον, να μπορεί να δώσει κίνητρα στην καινοτομία, αλλά αντιμετωπίζει και τα προβλήματα και του κινδύνου που αυτή η οικονομία που βασίζεται στην αξία των πληροφοριών να γίνει σωστά. Να γίνεται σωστή επεξεργασία των δεδομένων. Να αποφύγουμε τον κίνδυνο, όχι μόνο για την ιδιωτική ζωή, για την προστασία των δεδομένων που είναι πολύ σημαντικά, αλλά είναι και το θέμα τη ιδιοκτησία. Υπάρχουν διάφορε σημαντικέ στοιχείε νομικέ και θα τολμούσα να πω και διοντολογικέ, ηθικέ, που σχετίζονται με την ανάπτυξη, εξέλιξη τη ε, δημοκρατία. Άκουσα το πώ χρησιμοποιούνται τα δεδομένα κακώ αν δεν υπάρχουν σαφή κανόνε και να μην περιορίζεται η πρόοδο και η καινοτομία με στον κανόνα, αλλά θέλουμε πρόοδο και καινοτομία που θα εδράζονται επί τη προστασία των αξιών τη Ευρώπη. Να αποφύγουμε κινδύνου για τη δημοκρατία, με άλλα λόγια. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τωσενόφσκι έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αντιπρόεδρε τη Επιτροπή απρόσκοπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων έχει κέρια σημασία για την κοινωνία μας και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της διασφάλισης υποδομών που θα ανταποκρίνονται στις βέλτιστες προδιαγραφές. Η ταχύτητα μεταφοράς είναι μία προϋπόθεση, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ε, δυνατότητες ε, και τις υποδομές ε, χωρίς τις οποίες δεν θα μπορέσουμε να δράσουμε αποτελεσματικά. Αυτό έχει κέρια σημασία για τον δυναμικό χαρακτήρα των υπερδεδομένων των του τεράστιου δυναμικού που εμπλέκεται εδώ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια νέα προσέγγιση παράλληλη προς τα όσα έχουμε υιοθετήσει. Η ταχεία μεταφορά και οι υποδομές θέτουν ιδιαίτερες προκλήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε εκ του σύνεγγυς και να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες αποτελεσματικά. Ε, Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να έρθει το ψήφισμα στην Ολομέλεια. Στο μεταξύ, δίσαμε και την έκθεση για την ψηφιακή αγορά και για ξεκάθαρα λέμε τι θέλουμε για τα μαζικά δεδομένα. Το Κοινοβούλιο ξεκάθαρα ζήτησε να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον για την καινοτομία ε, στην ε, οικονομία που βασίζεται στα δεδομένα. Επίσης, ε, στην έκθεση ζητάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια διαφανή αξιολόγηση της κατάστασης για τα μαζικά δεδομένα. Δεν θέλουμε άλλη μελέτη, δεν είναι αυτός ο στόχος. Χρειάζεται μια επισκόπηση των πρακτέων, ούτως ώστε να τονώσουμε την καινοτομία και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που υπάρχουν, ε, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια οικονομία κλίμακα στην Ευρώπη. Μόνο έτσι μπορούμε να υποφεληθούμε από τα μαζικά δεδομένα. Δύο είναι τα ζητήματα που τίθενται. Πρώτον, η προστασία των δεδομένων και δεύτερον, δεξιότητες. Ας πάρουμε την προστασία των δεδομένων. Ελπίζω που τώρα υπάρχει, ε, σε σύντομα, συγγνώμη, θα υπάρξει το πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων θα προχωρήσει και με την πρωτοβουλία της ελεύθερης δροής δεδομένων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι χρειαζόμαστε απρόσκοπτη ροή, αλλιώς δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τις νέες τεχνολογίες που βασίζονται στα δεδομένα. Ε, και εμποδίζουμε την ε, ενιαία αγορά. Όμως δεν μιλάμε για προσωπικά δεδομένα, είναι, σε μεγάλες, ε, είναι μαζικά αυτά τα δεδομένα Και αυτά χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κλείσουμε συμπεράσματα και να τα χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις. Επίσης, όπως είπατε, κύριε Άνσιπ, μιλάμε και για δεδομένα που παράγονται από υπολογιστές αλλά από την άλλη όταν έχουμε τα μαζικά δεδομένα και κανένας δεν τα χρησιμοποιεί γιατί οι επιχειρήσεις δεν ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν, ε, τότε είναι άχρηστα. Περιμένουμε λοιπόν τις βασικές ε, κατευθυντήριες γραμμές για τις δεξιότητες για ε, στον τομέα αυτό. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γκραπίνη έχει μια γαλάζια κάρτα, κυρία Κάλλας. Τη δέχεστε? Ναι. Ωραία. Γκραπίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφε, στην ε, παρέμβασή σας ε, υποβάλλατε διάφορα ερωτήματα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το επιχειρήσεις επιχειρήσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε πως οι κανονισμοί που σχετίζονται με τα μαζικά δεδομένα λαμβάνουν υπόψη, τις επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη του Think Small First, ε, πρέπει να ρυθμίζουμε τα πάντα. Οι επιχειρήσει ε, παρότι δεν θα ταιριάζουν οι, νομοθετικέ οι νέες διατάξεις αυτές θα πρέπει να τι υιοθετήσουν παρόλα αυτά. Απάντηση. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Επειδή μιλάμε για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Ε, φυσικά θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και όταν προσπαθούμε να συζητήσουμε για του ε, κανονισμού των μαζικών δεδομένων, δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα μόνο τι μεγάλε επιχειρήσει, διότι σχεδιάζουμε τι διατάξει που τι βολεύουν εκείνε και όχι τι μικρομεσαίε στι επιχειρήσει και γι' αυτό χρειαζόμαστε χρόνο και ελπίζω να αφιερώσει τον πετούμενο χρόνο σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Ο κ. Ηλικιώτη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αξιοποίηση των νέων ψηφιακών δεδομένων πρέπει να έχει πρωταρχικό στόχο την ευημερία και την ενίσχυση τη ποιότητα ζωή των ανθρώπων. Δυστυχώ, σήμερα οι δυνατότητε τη τεχνολογία επιστρατεύονται για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολυεθνικών και του μεγάλου κεφαλαίου για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των επιχειρηματικών κερδών. γι' αυτό απαιτείται να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι και στο επίκεντρο να τεθούν οι ανάγκε και τα συμφέροντα τη κοινωνία. η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να προωθήσουν κρατικές επιδοτήσεις και δημόσιε επενδύσει για πλήρη αξιοποίηση των νέων ψηφιακών δεδομένων. στόχο πρέπει να είναι η πρόθεση τη έρευνα τη καινοτομία και τη ανάπτυξη η δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασία η διασφάλιση τη ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο η προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώ και η ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. εξίσου σημαντικό είναι να στηριχτούν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τεχνολογία για ενίσχυση τη θέση του στην αγορά και διευκόλυνση τη πρόσβαση του στη χρηματοδότηση. Mr. Helmer, ένα λεπτό. Πρόεδρε, 17 χρόνια είμαι εδώ στο Κοινοβούλιο. Ήμουν εδώ στο Συμβούλιο της Λισαβόνας ε, το Μάρτιο του 2000 και θυμάμαι τότε το στόχο που είχαμε θέσει να δημιουργήσουμε την ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία που βασίζεται στα δεδομένα μέχρι το 2010. Ε, όμως ε, οι μελέτες που θα γίνουν για την πρώτη δεκαετία του, αυτού του αιώνα θα δείξουν ότι η σχετική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχώρησε κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Όμως εμείς ε, συνεχίζουμε ε, ε ακάθεκτη και θέλουμε να φτιάξουμε μια θηρή οικονομία που βασίζεται στα δεδομένα. Ευτυχώ δεν έχουμε ε, συγκεκριμένο στόχο. Δεν θα ξέρουμε πότε έχουμε αποτύχει. Δεν μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από τι παρελθούσε αποτυχίε. Ε, έχουμε αυτές τις φοβερέ νομοθεσίε, ε, προσεκτικά επιλεγμένε λέξει. έρουμε τα εμπόδια, θέτουμε στόχο το επιχειρηματικό πνεύμα και την τόνωση τη βιομηχανία Καλό που την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπή να έχει ε, στο μυαλό της ακριβώς αυτό, να μην χρησιμοποιεί ε, την νομοθεσία για να επιτύχει τους στόχους τους, αλλά να ανοίξει επιτέλους τη στήριξη των νέων ευκαιριών. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κάμπελ, 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, για τα ε, ψηφιακά. Αν Κανένας ε, δεν μπορεί να θεωρήσει ότι παραμένει χωρίς να υποστεί τις επιπτώσεις ε, της ε, ψηφιακής αλλαγής. Ούτε καταναλωτής, ούτε, ούτε κράτη. Έχουμε επταπλάσια ταχύτητα από ότι ε, η αγορά αντιδρά και βλέπουμε εδώ ότι πρέπει να μπορέσουμε με τον καλύτερο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε ως Ευρώπη αυτές τις δυνατότητες. Οι ΙΠΑ βρίσκονται ως πρωτοπόροι πολύ μπροστά με πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Οι δυνατότητες που ανοίγονται είναι πολύ σχηδείς. Είτε πρόκειται για τις ε, νέες τεχνολογίες ε, και για τις δυνατότητες που διανοίγονται καθώς επίσης ε, και για τις, ε, τα αυτοκίνητα τα οποία με υπολογιστές μπορούν να κινούνται αυτόνομα. Βλέπουμε υπάρχουν και στην γεωργία ακόμα δυνατότητες όπου μηχανήματα μπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά και βλέπουμε εδώ και σε σχέση και με τα τρόφιμα και με το ε, νερό και την ε, δορυφορική υποστήριξη και όλες τις δυνατότητες που διανοίγονται. Τα μεγαδεδομένα ανοίγουν ε, μια νέα εποχή σε σχέση με τους, τις υπηρεσίες και τα ευφυή συστήματα μεταφορών. Κατά πόσον αυτό το δυναμικό θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε εξαρτάται από το βαθμό επενδύσεων και στις υποδομές και στην έρευνα και την ανάπτυξη. Έρευνα και ανάπτυξη καθώς επίσης και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα συνοδεύει αυτές τις ε, δραστηριότητες. Τα μέγα δεδομένα δημιουργούν ε, μια νέα κατάσταση στην Ευρώπη. Μέχρι το 2020 πρέπει να δραχθούμε της ευκαιρίας. Ευχαριστώ. Mr. Κύριος Κόρβιν Μίκε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Διαβάζω και βλέπω ότι χωλένουμε ίσως σε σχέση με άλλες χώρες που μας ε, έχουν υπερκεράσει, για παράδειγμα τι είπα, Ερωτώ, Κάποιοι συζητούν αυτά τα θέματα σε σχέση με το κοινοβουλευτικό επίπεδο για να μπορέσουν εταιρείε να δημιουργήσουν αυτά τα μεγαδεδομένα. Χρειάζονται όμως και ρυθμιστικά πλαίσια για τις δυνατότητες αυτές. Η αυταπάτη ότι εμείς δημιουργούμε αυτά τα μεγαδεδομένα είναι μια αυταπάτη. Καμιά χώρα δεν έχει κάνει κάτι ξεχωριστά. Όλες, ε, ε, όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και όλες οι πρόοδοι προέρχονται από από τις μεγάλες εταιρείες και όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε σχέση με αυτές τις βάσεις δεδομένων για τις πληροφορίες που χρειάζονται τηλεοπτικά ή διαφορετικά και πρέπει να θυμόμαστε ότι όλες αυτές οι πληροφορίες εκτός αυτών των μεγαδεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντικές υποθέσεις. Να μην αυτοφυλακιστούμε μέσα σε έναν αλαβάστρινο πύργο, ελεφάντινο πύργο. Θα πρέπει να δράσουμε πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ.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 Πρόεδρε, Επίτροπε, η αγορά των ονομαζικών δεδομένων είναι φυσικά μια ευκαιρία για την ανάπτυξη αλλά και πραγματικό κίνδυνο για του καταναλωτέ. Η γνωμοδότησή μου εστιάζεται σε τρία σημεία σε σχέση με αυτό το θέμα που έχουν ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να συνυπολογιστούν όταν υπολογίζουμε τα υπέρ και τα κατά. Πρώτον, είναι σημαντικό από τι μικρομεσαίε επιχειρήσει μέχρι τι πολυεθνικές να έχουν όλε οι επιχειρήσεις τι ίδιε ευκαιρίε να αποκομίσουν ωφέλη από αυτή την αγορά μαζικών δεδομένων. Ε, πρέπει να είναι ίση όροι ανταγωνισμού για να αποφύγουμε τα μονοπόλια όπω συχνά σήμερα στο τομέα τη πληροφορική ε, Δεύτερον, η χρήση των μαζικών δεδομένων ε, στι δημόσιε υπηρεσίε ε, Μπορούμε να διευκολύνουμε, να επιταχύνουμε την διοικητική διαδικασία, να δράξουμε την ευκαιρία για να καινοτομήσουμε και να είναι αποτελεσματικότερες δημόσιε υπηρεσίε. Τρίτον, και τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό σημείο, είναι μεγάλη η πρόκληση των μαζικών δεδομένων ω προ την προστασία των καταναλωτών. Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να αποφύγουμε τις εδόλες συμπεριφορές και τις ε, επιζήμιες για τους καταναλωτές ε, και παράτυπες συμπεριφορές. Ευχαριστούμε. Σαφχάουζερ, ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, με τις μεθόδους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, η μέθοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι, μας είναι εκεί. Υπάρχει ένα κέρδο και μας προβάλλουν όνειρα. Μας λένε, άμα τα κάνουμε όλα μαζί, θα έχετε περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερη παραγωγικότητα, περισσότερες θέσεις εργασίας. Όμως υπάρχει τελικά ε, ευρωπαϊκή στρατηγική, υπάρχει βούληση να έχουμε αυτόνομες πλατφόρμες όπως το Google, το Facebook, το Skype, υπάρχει βιομηχανική πολιτική ούτως ώστε να έχουμε ικανότητα, υπάρχει ικανότητα αποθήκευσης δεδομένων. Όχι είναι η απάντηση. Η ευρωπαϊκή στρατηγική είναι να ανοίξουμε ε, την πόρτα στις τεχνολογίες, αμερικανικές τεχνολογίες και στις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες που έχουν μονοπόλια για την επεξεργασία των μαζικών δεδομένων. Βασικό το πρόβλημα που θέλω να σε υποδείξω. Ε, η πρώτη ύλη είναι ο άνθρωπος. Ε, μήπω θα έπρεπε να απαγορεύσουμε ε, την χρήση αυτών των δεδομένων για μεταπόληση. Μήπω θα πρέπει να είναι η ιδιωτική ιδιοκτησία, η δημόσια ιδιοκτησία, αλλά θα πρέπει να είναι κοινοκτημοσύνη. Αυτή είναι, αυτό είναι το σύστημα που θα πρέπει να μα καθοδηγεί. Αυτό μπορεί να ισοδυναμεί με πραγματική ελευθερία. Ε, ευχαριστούμε κύριο Σχόκμαρκ Ε, πρόεδρε, πιστεύω είναι σημαντικό να τονίσουμε κάτι ότι η οικονομία που βασίζεται στα δεδομένα δεν είναι τίποτα καινούριο. Έχει ήδη παρέλθει αυτή η αλλαγή και Βλέπουμε στις οικονομίες ε, να υπάρχει με ε, μεγαλύτερη άνθηση εκεί που υπάρχει χρήση των νέων δεδομένων. Μην ε, μιλάμε για τα μαζικά δεδομένα σαν να είναι κάτι καινούριο, κάτι μαγικό. Ο στόχος θα πρέπει να είναι να βρούμε πώς θα τα επεξεργαστούμε τα δεδομένα, γιατί τα δεδομένα είναι γνώση και πρέπει να υπάρχει κατανομή και χρήση με νέους τρόπους ε, στην ε, σύγχρονη οικονομία. Και ο στόχος για μας θα πρέπει να είναι για την κυβερνοασφάλεια, για την ασφάλεια, για τη ροή των δεδομένων, ε, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα πνευματικά δικαιώματα, να καλύψουμε το κενό, να προσαρμοστούμε, να προσαρμοστεί η κοινωνία ώστε να μπορέσει να υποφελεί από τις ήδη φυστάμενες ε, δυνατότητες ε, που υπάρχουν. Με έναν τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα είμαστε οι καλύτεροι. Όπως είπε ο κύριος Σαφχάουζε και άλλοι, θεωρούν ότι είμαστε στο 19ο αιώνα ακόμη. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Μπορούμε να το αποφασίσουμε και να έχουμε ηγετικό ρόλο, να έχουμε την καλύτερη οπτική, είναι να έχουμε τις καλύτερες τεχνικές δυνατότητες και να δώσουμε τις δυνατότητες στην κοινωνία μας να είναι η καλύτερη. Μπορούμε να, να, να το αποφασίσουμε αυτό και αυτό θα πρέπει να κάνουμε, Πρόεδρε, κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ, κύριε Χακμάρ. Έχετε μια γαλάζια κάρτα από τον κύριο Ουζέλη. Τη δέχεστε? Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο εξή. Συμφωνώ βέβαια με αυτό το οποίο προαναφέρθηκε ότι πρέπει να προαχθεί η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις. Είναι σημαντική υπόθεση όμως οι Ευρωπαίοι πολίτες και για τους Ευρωπαίους πολίτες η προστασία των δεδομένων είναι το πιο σημαντικό θέμα και όχι μόνο για τα δεδομένα επιχειρήσεων που πρέπει να προστατεύονται, αλλά τα δεδομένα των πολιτών που πρέπει να προστατεύονται για την ιδιωτική του ζωή. Α σκεφτούμε για παράδειγμα τα θέματα των προσφύγων και τα συναφή προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά, πώς μπορούμε να δράσουμε ώστε να αντιμετωπιστούν απάτες, ε, πλαστογραφίες, ε, πλαστογράφηση και παρατυπίες σε όλους αυτούς τους τομείς. Ε, πρέπει να αναζητήσουμε μια νέα προσέγγιση πιστεύω εδώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ τα μάλα αυτή την ερώτηση, διότι μου δίνει την ευκαιρία να υπογραμμίσω και κάτι άλλο. Τα δεδομένα δεν είναι ένα μαγικό ψηφιακό θέμα, αλλά, δε, γνώση. Η γνώση έχει το χαρακτηριστικό ότι μπορεί να διανεμηθεί τάχιστα και να υποδιαιρεθεί επανειλημμένα. Μπορώ να σας δώσω γνώση, να μου δώσετε γνώση και πάλι θα έχουμε την ίδια γνώση πάνω μας. Αυτή είναι η μαγεία της γνώσης. Δεν αφορά τα στοιχεία, τα δεδομένα. Πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ. Τα περισσότερα δεδομένα Δημιουργούν το διαδίκτυο των πραγμάτων και το διαδίκτυο των πάντων, όχι τα προσωπικά δεδομένα. Αλλά στην οικονομία των δεδομένων μπορούμε να διαφυλάξουμε τα προσωπικά δεδομένα που θέλουμε να διαφυλάξουμε, αυξάνοντα ταυτόχρονα τα επίπεδα κυβερνοασφαλεία. Και σε γενικό ομαδοποιημένο επίπεδο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για έρευνα, επιστήμε, προστασία τη υγεία κλπ. Πολλοί από εκεί και από την άλλη πλευρά ίσω να μην το θέλουν αυτό. Εμείς όμως πιστεύω μπορούμε να καταλήξουμε σε συνεννόηση για τη χρήση των δεδομένων. Γνώση, διαφύλαξη ιδιωτική ζωής, αλλά και της ηγετικής θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόχρονα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κομπούλα Νάτρη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ψηφιακή οικονομία δεν έχει πολλά να προσφέρει. Ας δούμε τα γραφεία μας, ας δούμε τον εξοπλισμό μας, ας δούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν για ευρωπαϊκά προγράμματα και εξοπλισμό. Πρέπει η Ευρώπη να καταβάλει προσπάθειες, αλλιώς θα χάσουμε έναν της Ασίας και τον ΗΠΑ. Εμείς οι ίδιοι δεν θα παράξουμε τίποτα και θα χρησιμοποιούμε προϊόντα άλλων. Θα πρέπει να δούμε και όσον αφορά τις υποδομές να προαθούν οι εταιρείε και οι επιχειρήσει μα και να δούμε πώ μπορούν να διαδραματίσουν ένα ρόλο σε σχέση με του υπολογιστέ και την τεχνολογία. Όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τη δημιουργία μια εσωτερική ενιαία αγορα για τα ψηφιακά. Μια ψηφιακή αγορά και για την προσπάθεια προστασία των δεδομένων με νομοθεσία. Να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και κυρίω εναντί των καταναλωτών. Έχουμε ευκαιρίε ε, να γίνουμε ένα δραστήριος ε, που θα ε, παίκτης που θα συμμετέχει στα παγκοσμιοποιημένα αυτά θέματα και η προστασία αυτών των θεμάτων θα μπορέσει να είναι ένας γνώμονας για την Ευρώπη. Μπορούμε να δράσουμε αποτελεσματικά ως Ευρώπη και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, εκατομμύρια θέσεις εργασίας, αλλά πρέπει να δράσουμε σήμερα ήδη γι' αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, λέει Περνάμε μια πραγματικά συναρπαστική αρπαστική περίοδο. Από έναν πραγματικό κόσμο περνάμε σε έναν εικονικό κόσμο και τις δυνατότητες που διανοίγονται με αυτόν. Είναι μια μεγάλη πρόκληση να αναζητηθούν οι αλγόριθμοι και η μαθηματική βάση ώστε μέσα σε αυτό το νέο κόσμο να βρούμε ένα μπούσουλα, ένα μύτο της Αριάδνης ένα μύτο της Αριάδνης να πορευθούμε σωστά με τις καλύτερες βέλτιστες τεχνολογίες best enabling technology ώστε να παραμείνουμε πρωτοπόροι παγκόσμια και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή περίπου 200 δις ηλεκτρονικά μηνύματα διαχέονται καθημερινά βλέπουμε έναν όγκο δεδομένων που είναι αξιο, αξιόλογος. Έχουμε πάνω από ένα δις ε, στο facebook και έχουμε ολόκληρα δισεκατομμύρια και 2,6 δις ε, κινητά τηλέφωνα στην ε, παγκόσμια χρήση. Τα μπιτς που παράγονται είναι περισσότερα από τους κόκκους άμμου στις ακτές μας και τις παραλίες μας ε, και στις αμμουδιές μας ε, και έχουν διπλασιαστεί όλα αυτά μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο. Οι όγκη δεδομένων και η ανάλυση αυτών των δεδομένων και όλο το δυναμικό που υποκρύπτεται πίσω από αυτές τις δυνατότητες είναι τεράστιο. Πολλές θέσεις απασχόλησης και εργασίες μπορούν να δημιουργηθούν στο μέλλον. Με αυτή τη στρατηγική πρέπει γοργά να δραστηριοποιηθούμε, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Thank you. Ένα Ευχαριστώ. Μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω εστονικά και θα την αγράψω. Ε, θα ήθελα να πω πως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πάρα πολλά για να δημιουργήσει ένα δίκτυ της ε, ψηφιακής οικονομίας. Ε, δυστυχώς όμως ε, δεν είναι πολύ καλή εικόνα που αποκομίζουμε από τα δεδομένα φαίνεται ότι υπάρχει ένα χάσμα όταν ανάμεσα στα κράτη-μέλη Ιταλία, Ελλάδα, αν συγκριθούν ή και Βουλγαρία αν συγκριθούν με βόρειες χώρες, σκανδιναμικές χώρες, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ναι. χάσμα σε σχέση με τη χρήση των δεδομένων ή ακόμη και την χρήση του διαδικτύου. Χρειάζεται κατάρτιση, λοιπόν, εκπαίδευση, δεξιότητες για Ε, για, να, για την αρμοδιότητα των κρατών μελών για να επιταχύνουμε την διαδικασία χρειαζόμαστε κοινή προσέγγιση. Ε, όμως ε, ταυτόχρονα αν το αφήσουμε στα κράτη-μέλη δεν πρόκειται να προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα ούτως ώστε αυτή η οικονομία που βασίζεται στα δεδομένα να είναι το μέλλον της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ η ψηφιακή επεξεργασία των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στην έρευνα κλπ. Ε, είναι κάτι που αυξάνεται ανεφρηγουμένο. Από λίγα τεραμπάιτ του 2012 πήγαμε σε πολλά πέταμπάιτ σήμερα. Όπως ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, αυτή η εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει πολύ, πάρα πολλούς τομείς. Υγεία, ασφάλεια, ενέργεια, ε, συστήματα ευφυούς μεταφοράς και τεράστιο δυναμικό όμως οικονομικό για τις εταιρείε, δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξη νέων προτύπων επιχειρηματικών. Ο τομέας αυτός των Big Data δημιουργεί την ατότητα να εδραιωθεί στην πληροφορική η Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης. Γι' αυτό πρέπει να αρπάξουμε την ευκαιρία το ταχύτερο δυνατόν και να καλύψουμε το κενό που έχουμε τη ΣΥΠΑ. Για να δημιουργήσουμε λοιπόν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να ανθίσει η ενιαία αγορά των, ε, της μεγάλης μάζας δεδομένων πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει διελειτουργικότητα, προδιαγραφές, πρότυπα και να γίνουν επενδύσεις στο διαδίκτυο των πραγμάτων, ευρυζωνικές διασυνδέσεις της ταχύτητας, έρευνα, παιδεία, όλα αυτά πρέπει να προωθηθούν. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σόγκορ, δεχόσαστε μια γαντάζια κάρτα. κύριε Ρούμπικ. Uh, Μάλιστα. Ήθελα να ευχαριστήσω γιατί νομίζω επικεντρώνεται αυτό στο αναγκαίο σημείο. Με νέα ψαχτήρια νομίζετε ότι διανοίγονται νέες δυνατότητες για τους πολίτες και την ιδιωτική τους ζωή να μπορεί να, ε, να ε, εμπλέκεται. Πώς είναι δυνατόν ιδιαίτερα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, οικογενειακές επιχειρήσεις είναι μεγάλη πρόκληση να μπορέσουν να παρακολουθήσουν αυτές τις εξελίξεις νομίζω. Ευχαριστώ. Είναι αυτονόητο, ναι. Πιστεύω όμως ότι οι μικροί έχουν πάντα ένα μειονέκτημα δυστυχώς σε σχέση με τη μάχη που δίνουν να ανταγωνιστούν με τους μεγαλύτερους, τους ισχυρότερους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ευχαριστώ. So Ολοκληρώθηκε λοιπόν η παρέμβαση των πολιτικών ομάδων. Πάμε σε διαδικασία προσέγγισης προσοχής του Πρόεδρου. Η κυρία Βρέντα είναι η πρώτη που έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε τα μεγάλα, αυτά οι μεγάλοι μας δεδομένων, τα big data, μπορεί επηρεάσουν πολύ την κοινωνία θετικά, αν σεβαστούμε όμως την προστασία των δεδομένων. Και υπάρχει και μια ηθική διάσταση. Είναι σαφή. διότι άκουσα ανησυχητικέ ιδέε που εξέφρασαν κάποιοι συνάδελφοι για τον έλεγχο και τη διήθηση των προσφύγων, την ταυτοποίηση των ε, προσφύγων. Μπορεί να ωφεληθούν όλοι από τα θετικά στοιχεία και το δεδίκτυο για του πάντε και για τα πάντα Χρειάζεται. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται υποδομή ανοιχτή για την έρευνα και ισότιμη νομική προσέγγιση. Διάβασα στην Ανακοίνωση Ευρωπαϊκή για τα πνευματικά δικαιώματα με έκκληση μου ότι θα νομιμοποιήσει ε, την άντληση δεδομένων από, μόνο για δημόσιες υπηρεσίες έρευνας χωρίς να πληρώνονται πνευματικά δικαιώματα. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε πολύ τα δεδομένα αυτά, αν οι καινοτόμες εταιρείες, οι πολίτες και επιστημονικά προγράμματα αντιμετωπίζουν νομική αβεβαιότητα όσον αφορά ε, τον ξεπερασμένο νόμο για πνευματικά δικαιώματα. Από τη μία πλευρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι χρειάζεται σύμπραξη του ιδιωτικού δημόσιου τομέα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα. Ταυτόχρονα όμω, από την άλλη, η συμμόρφωση στου του κανόνε πνευματική ιδιοκτησία δεν είναι δυνατόν για προγράμματα που χρησιμοποιούν τα big data με τη συμμετοχή του δημόσιου τομέα. Πρέπει να, αντλούνται, να αντλείται περιεχόμενο από διάφορου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων που είναι χιλιάδε εκατομμύρια. Χρειάζεται απλούστευση των κανόνων περί πνευματική ιδιοκτησία για όλου του φορεί, εμπορικού, μη εμπορικού. Μόνο έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τι δυνατότητε που προσφέρονται και τα πνευματικά δικαιώματα να μην αποτελέσουν τελικά εμπόδιο την ανάπτυξη του τομέα αυτού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πολτσέκ είναι ο επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε πολλές τυχές αναφέρθηκαν όσον αφορά την οικονομία των μεγαδεδομένων ιδιαίτερα και με τα ιδιωτικά δεδομένα και την προστασία τους προστασία επίσης επιχειρησιακών δεδομένων προστασία ε, δικαιωμάτων ε, πνευματικής ιδιοκτησίας και όλα αυτά σε ένα ε, ευέλικτο ελαστικό πλαίσιο. Υπάρχει και ένα θέμα εδώ, copyright, πνευματικά δικαιώματα έναντι της ταχείας συνένεσης ε, για την χρήση δικαιωμάτων, πνευματικών δικαιωμάτων. Η ταχύτητα εδώ όσον αφορά την συνένεση που απαιτείται για την χρήση τέτοιων δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ σημαντική πτυχή και θα έλεγα, θα προσέθετα ότι είναι ένα ευάλωτο στοιχείο, ένα τροτό σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν έχουμε μια κοινή ενιαία αγορά ε, εφόλων αυτών και έχουμε πολλά προσκόμματα και εμπόδια ακόμα. Ευχαριστώ. Uh, Ο Καπούτο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνέταξα πάρα πολλέ ερωτήσει, παρεμβάσει και δηλώσει όσον αφορά την ανάπτυξη διαδικτύου και όσον αφορά την χρήση των big data για τον εξυγχρονισμό τη οικονομία και τη δημόσια υγεία. Υπογράμμισα όμω και την άλλη όψη, δηλαδή το Wi-Fi που ακτινοβολεί, ε, τη κυκλοφορία, τις απάτε στον τομέα τη πληροφορική, το λαθρεμπόριο των φαρμάκων. Είναι πρόκληση οι καθολικέ υπηρεσίε του διαδικτύου για να έχουμε σωστέ υπηρεσίε Καθολική όπω την ηλεκτρονική υγεία. Χρειάζεται σωστή θάθμιση, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων, μεγάλο σοβασμό τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Μόνο κανόνε καθορισμένοι δημιουργούν θετικό αντίκτυπο πολιτισμικό και κοινωνικό. Δημιουργούν ενιαία αγορά ψηφιακή, μισότιμε συνθήκε στι επιχειρήσει και ασφάλεια για του πολίτε. Συμφωνώ με την ερώτηση και προσθέτω ότι πριν από τι μέρε είπατε εκπρόσωπο του ΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ζαΐντ Ουσέιν, είπε στη ΣΥΠΑ πρέπει να χωρίσουν πολύ προσεκτικά όσον αφορά το θέμα της Apple με την FBI, τη διαμάχη. Γιατί μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στα ανθρώπινα δικαιώματα για όλο τον κόσμο αυτή η διαμάχη. Ποια απάντηση μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα της διαμάχης Apple-FBI. Ο κύριος Μαριάς, ο τελευταίος που έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε επισημάνει πολλάκις ότι τα κονδύλια που έχουν επενδυθεί στον τομέα των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολείπονται των επενδύσεων που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιαπωνία. Ωστόσο η κάλυψη της απόστασης δεν πρέπει να στηρίζεται στην κινεζοποίηση των μισθών και των συνθηκών εργασίας. Σίγουρα η ευρωπαϊκή νομοθεσία οφείλει να προσαρμοστεί στη διασυνοριακή αρχιτεκτονική του διαδικτύου ώστε να γεφυρώσει τις διαφορές τη κατακαιρματισμένη Ευρωπαϊκή Αγορά. οφείλει όμω να προστατεύσει και του πολίτε των κρατών μελών. γι' αυτό θα πρέπει να σταματήσει η περαιτέρω απελευθέρωση τη αγορά, ιδίω στον τομέα των υπηρεσιών που επιχειρείται με την tisa. με άλλα λόγια η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει εκτό των άλλων να αναγνωρίσει και να προτείνει ένα σαφέ πλαίσιο αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση τη οικονομία για του εργαζόμενου, τόσο όσον αφορά τι θέσει εργασία όσο και την ψυχική και σωματική του υγεία μεριμνώντας για την προσβασιμότητα των πολιτών στο διαδίκτυο θέματα που δεν θίγονται στην προφορική ερώτηση. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώνεται η διαδικασία και για να ολοκληρωθεί και η συζήτηση ο Αντιπρόεδρος Άνσιτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ και πάλι για τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί να μεγιστοποιήσει το μεγάλο δυναμικό των δεδομένων υπέρ της οικονομίας σε μια ενιαία στρατηγική για την εσωτερική αγορά και άλλες δράσεις της. Συμφωνώ με την κυρία Βίκη Φόρντ, Ευρωβουλευτή η οποία προανέφερε ότι τόνισε τη σπουδαιότητα ώστε στις ε, ηλεκτρονικές ε, συμβάσεις ε, να χρησιμοποιούμε αυτή τη δυνατότητα. Ο κώδικας και των διαδικασιών για την χρήση αυτής της δυνατότητας ηλεκτρονικά μπορεί να δώσει 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετήσια μεγάλο ποσό και δυστυχώς δεν έχουμε ένα τέτοιο ποσό στη διάθεσή μας. Πρέπει να εισαχθούν σε όλα τα κράτη-μέλη ηλεκτρονικοί λογαριασμοί και η δυνατότητα ηλεκτρονικών υπογραφών για εξοφλήσεις θα πρέπει να προστατεύσουμε τον, την ιδιωτική σφαίρα των πολιτών μας σε σχέση με τα ιδιωτικά τους προσωπικά δεδομένα τα κοινοβούλια, πρέπει να ανοίξουν τα δεδομένα τους σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλες τις συνιστώσεις και συντελεστές, ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι σημαντική υπόθεση για αυτές, αλλά και για τους μεγαλύτερους παίκτες που εμπλέκονται. Το ψηφιακό ζήτημα έχει μεγάλη σπουδαιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό όχι μόνο σε σχέση με τα κράτη-μέλη αλλά και στα ίδια τα κράτη-μέλη και σε εκείνα τα κράτη-μέλη όπου η τεχνολογία των πληροφοριών έχει αναπτυχθεί σε ανώτατο επίπεδο μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ένα χάσμα ηλεκτρονικό και ψηφιακό μεταξύ των αστικών κέντρων και των ε, περιοχών της Υπέθρου, μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων, των γυναικών ε, και των υπόλοιπων ε, μελών του πληθυσμού μας μου δώσατε ένα λεπτό και έχω χρησιμοποιήσει ήδη, έχω αναλώσει δυόμιση λεπτά. Λυπούμε που δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει νομοθετικά όλα αυτά με προτάσεις της σε όλα αυτά τα θέματα το επόμενο έτος θα πρέπει να δράσουμε με ιδιαίτερη ταχύτητα να επιτύχουμε τους ρυθμούς μας φυσικά και στρέφομαι προς εμάς ο κίνδυνος είναι να χάσουμε στον ανταγωνισμό αυτό ως Ευρώπη έναντι άλλων εμπλεκόμενων. Και γι' αυτό πρέπει να βιαστούμε, να επιταχύνουμε τις διεργασίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. Προσβλέπω στο να μπορέσουμε με τους συνομοθέτες γοργά να δράσουμε και να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις για την οικονομία που θα βασίζεται στα δεδομένα και θα αποτελέσει δυνατότητα να αποβεί προς όφελος όλων του ιδιωτικού τομέα και των πολιτικών πολιτών και των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε εμείς, Αντιπρόεδρε. Κλείνει η συζήτηση.